Dear colleagues, we can continue. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το 9 που το έχουμε αφήσει το πρωί. Ο λόγος στην κυρία Λεκρύπ. Πρόεδρε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσον αφορά το θέμα των ψηφιακών πλατφορμών. Σημαντικό θέμα. Και λίγο ακόμη για τον ορισμό, την ομασία των πλατφορμών αυτών. Το έχουμε συζητήσει επαρκώ το θέμα. Συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για τεράστιο θέμα. Είναι πολλά τα διακυβεύματα εδώ, πολλές ανησυχίε, πολλές οι απόψει. άπτεται άλλωστε πολλών άλλων θεμάτων που συζητούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Εμείς ε, ως Επιτροπή Γιούρι εξετάζουμε έκθεση πρωτοβουλίας που συντάσσουν από κοινού οι Ήτρε και η ΙΜΚΟ. Εμείς γνωμοδοτούμε μετά και υπό το φως της ανακοίνωσης περί τον Μάιο, ανακοίνωση της Επιτροπής για τις προκλήσεις ε, που άπτονται των ψηφιακών πλατφορμών. Μεταξύ αυτών έχουμε και το θέμα της ευθύνης αυτών των ψηφιακών πλατφορμών. Τεράστιο θέμα Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σκεφτούμε. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο, ούτε καν ε, σήμερα. Και, και δι σήμερα θα έλεγα, λόγω του κοινοβουλευτικού έργου. Εν πάση περιπτώσει εμείς απλώς γνωμοδοτούμε, η Ήτρε και η ΕΜ, ΙΜΚΟ πάντως θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα. Δεδομένου συνεπώς του περιορισμένου χρόνου, και επειδή πρέπει να γνωμοδοτήσουμε επί εκθέσεω πρωτοβουλία, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το κείμενό μου είναι καταρχάς σύντομο. Μία σελίδα μόνο, στο οποίο επιδερμικά και μόνο πραγματεύουμε κάποιες βασικές πτυχές του θέματος. Ελπίζω ότι κατάφερα να καλύψω τις περισσότερες βασικές πτυχές του θέματος εκ μέρους της Επιτροπής Γιούρη. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα θελήσει να πει δύο λόγια για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι μας αφορά εναντί λοιπόν των δύο άλλων επιτροπών. Ε, το θέμα είναι ο ορισμός. Τι σημαίνει ψηφιακή πλατφόρμα. Πιστεύω ότι πρόκειται για προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε καλή νομοθεσία. Η ποικιλία των πλατφορμών και των δραστηριοτήτων τους είναι τέτοια που είναι σκόπιμο να δοθεί ένας ακριβής πλήρης ορισμός των πλατφορμών και των δραστηριοτήτων τους. Όσον αφορά το θέμα της ευθύνης, επικεντρώθηκα σε αυτήν την σύντομη γνωμοδότηση επί του θέματος που άπτεται περισσότερο του αντικειμένου της Επιτροπής μας συγκεκριμένα ευθύνη έναντι των πνευματικών δικαιωμάτων. Και λίγα σχόλια για το εμπορικό δίκαιο, τα δικαιώματα των επιχειρήσεων κλπ. Οι πλατφόρμες αυτές λοιπόν φέρουν ευθύνη εναντί των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και ε, για την διαφάνεια και την πίστη που οφείλουν στους πελάτες τους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους Υπνομικού χαρακτήρα, βιομηχανικού κλπ. Οι πλατφόρμες αυτές είναι εξαιρετικά ισχυρές εναντί πολλών άλλων παικτών. Επικεντρώνομαι λοιπόν σε αυτές τις πτυχές που από τον όπως είπα του αντικειμένου της Επιτροπής μας υπάρχουν και άλλες πτυχές που αφορούν τις πλατφόρμες αλλά για τα άλλα εμές τις δύο καθήλυν αρμόδιες επιτροπές. Γιατί όπως προείπα το θέμα είναι τεράστιο. Εμείς πιεζόμαστε χρονικά, άρα ας προσπαθήσουμε σήμερα να πούμε δύο λόγια και να κλείσουμε. Να θέσουμε και μια προθεσμία θέση τροπολογιών. Θα είναι πολύ κοντινή γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ταχύτερα. Η προθεσμία αυτή είναι αρχή επόμενης εβδομάδας. Δευτέρα 27 Μαρτίου. Δευτέρα 27 Μαρτίου. Είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει επιδέξιους χειρισμούς για να μπορέσουν οι δύο καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές να ψηφίσουν στις επόμενες συνεδριάσεις τους. 11 και 12 Απριλίου συγκεκριμένα. Προκαταβολικά λοιπόν, συγγνώμη για την πίεση, αλλά έτσι τα πράγματα. Έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις. Πρόεδρε, είδου το κείμενό μου. Ε, δεν μου άρεσε και το ότι έπρεπε να είμαι τόσο σύντομη. Θα χρειαστεί ενδεχομένω να καταθέσω και αυτοτροπολογίες, τροπολογίες επί του κειμένου μου, γιατί κάποιες διορθώσεις θα χρειαστούν. Όπως είπα, έπρεπε να κάνω ότι έκανα υπό μεγάλη χρονική πίεση. Αυτά προσβλέπω σε μια καλή συζήτηση. Κύριε Ρέγκνερ. Πρόεδρε. Διαβάζω την άποψη του κ. Κοφεράτη, ο οποίος δεν Ευχαριστεί την κυρία Λεγκρίπ, βεβαίως. Οι πλατφόρμες χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τη ζωή του Ευρωπαίου πολίτη. Έχει μεγάλη σημασία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συζητήσουν τον ρόλο τους μαζί με τους ε, αρμόδιους φορείς. Το θέμα είναι τεράστιο, εννοείται πέραν των νομικών πτυχών. Έχει μεγάλη σημασία όμως να είμαστε παρόντες σε αυτήν την συζήτηση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλιώς η κάθε χώρα θα κάνει τα δικά της, ενώ το θέμα είναι να κάνουμε κάτι ως Ευρώπη. Και Σκοφέρα, θα ήθελε να επιμείνουμε επί του ορισμού. Παρακολουθεί τη συζήτηση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ευρύτατο πλαίσιο. Ο ορισμός να είναι λοιπόν αρκετά γενικός. Για την Επιτροπή μας το θέμα της ευθύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ζωτική σημασία να διατυπώσουμε με σαφήνεια τους κανόνες ευθύνης. Οι πλατφόρμες είναι ενδιάμεση ή δεν είναι για παράδειγμα μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει και εδώ. Και υπάρχουν και άλλες πτυχές που θέλει να τονίσουμε. Φορολογία. Όλοι γνωρίζουμε το θέμα, όχι μόνο μέσα των Panama Papers, αλλά και μέσα των LuxLeaks. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Πώς παρακολουθούνται οι συναλλαγές, οι σχέσεις επασχόλησης, οι συνθήκες εργασίας που συζητήθηκαν ήδη στην Επιτροπή Επασχόλησης. Υπάρχει λοιπόν και μια κοινωνική διάσταση. Να μην ξεχάσουμε τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές, τις συνθήκες εργασίας όπως προείπα και δύο άλλα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε ε, και το θέμα της φορητότητας να το συζητήσουμε οι χρήστες πλατφορμών που ενδιαφέρονται για την φορητότητα και ο κύριος Κοφεράτη επίσης θέλει να δούμε το θέμα των ε, πλέον ευάλωτων ομάδων μεταξύ αυτών και τα παιδιά που εκτίθενται υπερβολικά σε μηνύματα σεξιστικά και άλλα. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να δεσμευθούν για την προστασία των ευάλωτων αυτών ομάδων. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα. Ε, φυσικά προσβλέπουμε σε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Α, κυρία ζητήσε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγητή για το σχέδιο συζητάμε μια παλιά ανακοίνωση, δηλαδή του Μάη του 16. Για να έχουμε λοιπόν προσθέμενη αξία στη δουλειά μας εδώ, πρέπει να επικεντρωθούμε στις πρωτοβουλίες της ανακοίνωσης για τις πλατφόρμες, όπου ακόμα η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση νομοθεσίας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ανδέλφους που εργάζονται σε αντίστοιχους φακέλους και πρέπει επίσης να με υπόψη μας θέματα όπως δίκαιες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, διαφάνεια, διαλειτουργικότητα, σημαντικά θέματα για μας όσον αφορά τη μετάβαση από μια πλατφόρμα σε άλλη και αλλαγή υπηρεσία. Βέβαια, εδώ στο επίκεντρο είναι το θέμα της λειτουργικότητα και μεταξύ πλατφόρμων. Βέβαια, εδώ όταν μιλάμε για πλατφόρμες έχουμε κάποιον διάμεσο. Κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια έχουμε και ένα καθεστώς περιορισμένης ευθύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και εμεί λέγαμε πάντοτε ας πούμε στην ε, μεταρρύθμιση ψηφιακής αγοράς ότι θα πρέπει να προσέξουμε γιατί για τις πλατφόρμες όπως Spotify και Netflix να δούμε τι γίνεται γιατί δεν είναι διάμεση. Οπότε πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο και να είμαστε προσεκτικοί ώστε να εφαρμόσουμε την τωρινή, την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και όχι να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Αλλιώς θα δημιουργήσουμε πολύ ανασφάλεια δικαίου γιατί και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο διασφαλίζει νομίζω σημαντική προστασία και θεμελιώδη δικαιώματα στα πλαίσια της καινοτομίας. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο ως επόμενο βήμα από την Κομισιόν να προτείνουμε μία διευκρίνηση ή αποσαφήνιση για το πώς ακριβώς αφαιρούν οι διάφορες πλατφόρμες το παράνομο ή μη λοιπόν πρέπον περιεχόμενο. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υπάρχει μια ιδιωτική εφαρμογή δικαίου. Να αποφασίσει δηλαδή τι επιτρέπεται κανείς και τι δεν επιτρέπεται μόνος του. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές, το τι πρέπει να αφαιρούν και πόσο σύντομα και πρέπει να έχουμε καλύτερες πληροφορίες προς αυτούς που υποβάλλουν αυτά τα αιτήματα, πώς θα πρέπει να και κλπ. Λέει η Κομισιόν θα πρέπει να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά, παρά να αλλάξουμε εκ βάθρων, δηλαδή την ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευχαριστώ κύριο Καβαντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα να πω στην κυρία Λεγκρίπ ότι συμφωνώ εδώ με αυτά που είπατε και στηρίζω απόλυτα το περιεχόμενο των θέσεών σας ξεκάθαρα και μετάκλητα δεν χρειάζεται λοιπόν μια και συμφωνώ εφόλου λύση να σας πω επί ποιον θεμάτων συγκεκριμένα συμφωνώ ευχαριστώ η Κομισιόν επιθυμεί το λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ. Από την Γενική Διεύθυνση Connect της Επιτροπής. Ευχαριστώ για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Θα τα πω σύντομα. Παρατηρήσεις. Για αυτό το σχέδιο. Εμεί καλωσορίζουμε τη συζήτηση και όπως είδατε κι εσείς κάνουμε κάποια δουλειά πάνω στους ορισμούς και ήδη έχουμε συνοδευτικά έγγραφα για τους ορισμούς ώστε να καθορίσουμε το τι αποτελεί πλατφόρμα και κατά πόσο θα ήταν καλό να δώσουμε ένα ενιαίο ορισμό πλατφόρμας, τη στιγμή που υπάρχουν διάφορες, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδο. Αντί λοιπόν να δώσουμε έναν ιόρισμό, ίσως να ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ πλατφορμών. Και αυτό είναι και η βάση πάνω στην οποία δουλεύουμε εμείς. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η πολύπλευρη φύση αυτών των πλατφορμών και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν. Συχνά προσωπικά. Στόχος μας στην πολιτική ήταν να διασφαλίσουμε ένα υγιές οικοσύστημα οικονομίας πλατφορμών και όχι μόνο να κρίνουμε αν έχουν αρνητικό θετικό ρόλο οι πλατφόρμες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα οικοσύστημα υγιές λοιπόν, όπου οι πλατφόρμες θα διευκολύνονται να βρουν ένα ρόλο ιδιαίτερα για τις μικρές και μικρές κεφαλαιοποίησεις πλατφόρμες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στο 4% που αφορά δηλαδή τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες παγκοσμίω. Αυτό βέβαια είναι μια οικονομική δυναμία στα πλαίσια της οικονομίας των πλατφορμών. Και το δυναμικό καινοτομίας πάντως των πλατφορμών από την Ευρώπη είναι ισχυρό. Το κείμενο τώρα που προτείνει η συγγετρία το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και να σας πω ότι όπως προείπαν κι άλλοι για τα πραγματικά δικαιώματα ήδη έχουμε συγκεκριμένε νομοθετικές προτάσεις από την Κομισιόν οπότε καλύτερα να το εξετάσουμε σε αυτό το πλαίσιο και όχι στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για τις online πλατφόρμες. Και ευχαρίστω να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αν χρειάζεται. Μας ενδιαφέρει επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα την, το θέμα της διαφάνειας, της ε, συχνής ε, παρουσίας των πελατών και ε, όπως είπε και κάποιος, τι γίνεται με τις κοινοποιήσεις για την ανάρτηση και κατέβασμα περιεχομένου. Αυτά πάντως από μένα. Να ευχαριστήσω και πάλι την συγκήτρια και ευχαρίστω να σας δώσω οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια επιθυμείτε όποτε το κρίνετε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα, λέει ο Πρόεδρος και να συνεχίσουμε με το σημείο 10. Αναλογία απόψεων για τους κανόνες που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Ο κύριος ε, Βόλκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από πολλές διαβουλεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατέθεσε τις νομοθετικές της προτάσεις για την ψηφιακή αγορά. Ε, και επίσης και για τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Καταρχήν, όσον αφορά τη διαδικασία, τόσο η Επιτροπή ΙΜΚΟ όσο και η Επιτροπή ΚΟΥΛΤ ε, κατέθεσαν σχέδιο της γνωμοδότησής τους. Ε, η ΚΟΥΛΤ συμμετέχει στο άρθρο 55 και η γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο. Επί της ουσίας, ε, δεν θέλω να σπαταλήσω πολύ χρόνο. Ε, θα ήθελα με μεγάλη χαρά να ακούσω τις ε, απόψεις των σκιωδών. Και βεβαίως ε, θα ήθελα ή θέλω να πω ότι γνωρίζω ότι το θέμα είναι επίμαχο. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ το βήμα που θέλουμε να κάνουμε είναι σωστό. Ο κανονισμός αναφέρεται στον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ψυχαγωγικές επιτροπές για τους πολίτες. Όμως σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει περιορισμός και έτσι συγκεκριμένα από 122 τηλεοπτικά κανάλια στην Πολωνία μόνο δύο μπορούν να ληφθούν στη Δανία. Ε, τα πράγματα λοιπόν είναι αρκετά δυσάριστα. Το 82% των ε, τηλεοπτικών σταθμών και το 62% των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών ε, χρησιμοποιούν το geo-blocking. Παραδείγματο χάρη, ένα ε, τσεχικό σταθμό μπλοκάρει το σύνολο του προγράμματό του. Κατά την άποψή μου, η πρόταση που έχει κατατεθεί, η πρόταση αυτή μπορεί τελικά να οδηγήσει ε, κοινή αγορά στο ψηφιακό τομέα. Στις διαβολεύσεις που είχα, ε, ετέθη ένα αμφιβόλιο ο στόχος αυτής της ε, πρότασης και εδώ θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Με τον κανονισμό της κινητικότητας, το Slack Flexi Sky Snack, ε, στο μέλλον θα μπορούν όλα αυτά να είναι διασυνοριακά, όμως για περιορισμένη διάρκεια. Ο κανονισμός ως εκ τούτου ρυθμίζει μόνο τις υπηρεσίες εκείνες που έχουν αγοράσει οι πολίτες με το CapSat Online, οι πολίτες ανεξάρτητα από την πικότητά τους και τον χώρο εγκατάστασής τους. Αυτοί έχουν κάποια πρόσβαση και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο Netflix, αυτό έχει κοινωνική διάσταση. Μπορούν να υποφεληθούν κυρίως οι γλωσσικές μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπρόσθετα 15 εκατομμύρια άνθρωποι οποίοι ε, μπορούν να εκμεταλλευτούν την κινητικότητα και να εργάζονται σε άλλη χώρα. Επιπλέον η Ευρώπη σε παραμεθόριες περιοχές θα γίνει πολύ ζωντανή και θα δώσει τη δυνατότητα ε, οι άνθρωποι να απαλλαγούν από τις παλαιότερες τεχνολογίες ε, ε, κάποιας γειτονικής χώρας, να μπορούν να περάσουν στις νέες τεχνολογίες. Η δική μας η πρόταση προτείνει έτσι ώστε κυρίως τα ψυχαγωγικά προγράμματα και ειδήσει να είναι πιο εύκολα προσπελάσιμα και κυρίως ε, σε μια εποχή των δαϊκίστικων ειδήσεων να υπάρχει καλύτερη ποιότητα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μισό λεπτό πραγματικά ειλικρινά μιλάτε με τέτοια ταχύτητα. Αυτή είναι ταχύτητα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 σε μια κοινωνία της πληροφορίας υπάρχουν ε, σημαντικές ε, πληροφορίες οι οποίες ε, προσφέρονται από κλασικούς φορείς και πολλές υπηρεσίες δεν μπορούν να αγοραστούν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στη δημοκρατία μας και επιπλέον και αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε αλλάζει και η συμπεριφορά των θεατών. Όλο και πιο νέοι βλέπουν προγράμματα online άρα δηλαδή στην νομοθεσία θα πρέπει να γίνεται κάτι για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Σήμερα είδαμε ήδη στις επιγραμμικές ε, ανταλλαγές ότι αυτά είναι όλο και πιο σημαντικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ ε, σημαντικό να μην αγνοήσουμε τις επιγραμμικές ε, αγορές και σήμερα να μην δίνουμε δυνατότητα σε γκρίζες αγορές και Θεωρώ ότι θα πρέπει τις εκπομπές να τις αγοράζουμε, να πληρώνουν οι άνθρωποι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, αυτά τα χρήματα, ε, να μην τα τοποθετούμε σε VPN, τέτοιου είδου ε, δοσολογίες, αλλά να βάλουμε εμπόδιο στην πειρατεία. Και τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο του κανονισμού, ο κανονισμός αυτός αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Το άρθρο 2 αναφέρει την αρχή της χώρας προέλευση ε, και καθορίζει ότι η ραδιοτηλεπτική παραγωγή ε, θα πρέπει να σέβονται μόνο το δικαίωμα του δημιουργού από τη χώρα όπου γίνεται η ε, μετάδοση. Επίσης θέλω να πω, αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι πρώτον η ελευθερία ε, των συμβάσεων και δεύτερον ε, το ε, δίκαιο της κάθε χώρας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Κυρίως αυτό μερικές φορές το λένε πολλοί, κυρίως δεν θα υπάρξει πανευρωπαϊκή άδεια, αλλά ο κανονισμός επιτρέπει σε τηλεοπτικούς σταθμούς να ασκούν ε, μόνο κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα και πρέπει να πούμε με σαφήνεια. Παρά αυτές ε, τις απλουστευμένες διαδικασίες ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις άδειε το πόσο μεγάλο είναι το κοινό και εδώ θα ήθελα να προτείνω καλύτερη διατύπωση Τέλος λοιπόν, θέλω να πω ότι ως digital native ε, επιτιμώ να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και λόγω του ότι ε, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, ε, είμαι αρκετά επιφυλακτικός γιατί για να υπάρξουν ε, αλλαγές χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Να πω κάτι, ελπίζω κάποιοι να τοποθετηθούν από αυτού. Υπάρχουν οι ανησυχίες των παραγωγών, εκφράστηκαν αυτές οι ανησυχίες και τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου. Και αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον κινηματογράφο στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Από την άλλη όμως δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι η επέκταση στον επιγραμμικό τομέα πράγματι θα καταστρέψει το επιχειρηματικό μοντέλο αυτής της ομάδας ε, διότι υπάρχουν γλωσσικοί φραγμοί ε, και εκτός αυτού εξακολουθεί να ισχύει η ελευθερία των συμβάσεων. Αυτά είχα να σας πω και χαίρομαι που θα ακούσω ε, τις ερωτήσεις που, την κυρία που μόλις τώρα από τη συνάδελφη που μόλις μπήκε στην έρευνα. Ε, Ευχαριστώ κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά που είπε. Εγώ Είμαι αρμόδια για τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών. Σε πολλά θέματα συμφωνώ. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και αυτή η οδηγία σε τελική ανάλυση είναι ένα κάποιο βήμα προς την κατεύθυνση της διασυνοριακής ε, πρόσβασης ε, σε εκπομπές. Η Κομισιόν είχε πει ότι θα καταργήσει το geo-blocking, ότι είναι διακριτική μεταχείριση, σήμερα πια όμως δεν το λέει πια αυτό. Και πολλές ανησυχίες ε, που είχαν εκφράσει οι δικαιούχοι δικαιωμάτων, αυτές οι οδηγίες είχαν αναφερθεί και αρχές της δεκαετίας του 80 για το ZATCAP και τότε όμως παρόλα αυτά στην πράξη αποδείχθηκε ότι είναι καλή αρχή της χώρας προέλευσης και με τον τρόπο αυτό οι γλωσσικές μειονότητες στις παραμεθόριες περιοχές είναι σαφές ότι θα μπορούν να έχουν λήψη εκπομπών στη μητρική τους γλώσσα. Ε, στο ίντερνετ όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτή είναι μια αδικία η οποία σε τελική ανάλυση οδηγεί στο ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή από το να ε, βλέπουν εκπομπές παράνομα διότι το geo ιδιαίτερα σε ραδιοφωνία ραδιοφωνικές εκπομπές όπως είναι τα ε, ντοκιμαντέρ. Ε, ε, αυτά δεν μπορούν να προστατευτούν και σε άλλες χώρες βέβαια δεν έχουν και καμία χρήση. Εγώ την πρόταση της Επιτροπής τη βρίσκω καλή και θέλω να πω όσον αφορά την ελευθερία των συμβάσεων ότι προφανώς και δεν αλλάζει τίποτα στην ελευθερία των συμβάσεων με την αρχή της χώρας προέλευσης. Παρόλα αυτά ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τις ε, διατάξεις της οδηγίας ε, για την δορυφορική και την καλωδιακή τηλεόραση τότε η ίδια η Κομισιόν είχε πει ότι η ελευθερία των συμβάσεων είναι η αχίλιο επτέρνα αυτή τη οδηγία και για το λόγο αυτό ε, σε πολλέ ε, δορυφορικέ εκπομπές υπάρχουν πράγματα που δεν μεταδίδονται. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι και η συμβασιακή ελευθερία έχει όρια κυρίως όταν πρόκειται για ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ως προ την αρχή της χώρα προέλευση, νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές ότι η ίδια η αρχή αυτή ρυθμίζει το ε, πιο δίκαιο ε, δημιουργού ισχύει και που όχι και όχι το τι περιλαμβάνει, το, το περιεχόμενο δηλαδή μιας άδειας. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να φορέσουμε κορσέ στις ε, εκπομπές ε, γιατί σε τελική ανάλυση όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και με τα επίκαιρα τηλεοπτικά προγράμματα. Εγώ θεωρώ ότι ε, αυτή η αρχή της χώρας προέλευσης είναι αποδεκτή για τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Τώρα, όσον αφορά τους, ε, τα συγκεκριμένα δικαιώματα για την ε, περαιτέρω αναμετάδοση. Εδώ ε, δεν έχει καμία σημασία κατά πόσον η αναμετάδοση θα γίνεται μέσα από ένα κλειστό δίκτυο ή από το διαδίκτυο. αυτό που κάνει τη διαφορά είναι αν χρειάζεται κάποιο password ή όχι. Είναι σημαντικό να γίνονται όλα αυτά και μέσα από το διαδίκτυο γιατί ο κανονισμός φορητότητας που θα ε, ψηφίσουμε αύριο μπορεί να ε, είναι εφικτός μόνο όταν και μια εκπομπή είναι φορητή. Γιατί αν κάτι ε, δεν μπορεί να μεταδοθεί από το διαδίκτυο, κατ' ουσίαν αφαιρούμε πολλά στοιχεία από την αρχή της ε, φορητότητας. Και σε τελική ανάλυση είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει θέματα που έχουν ρυθμιστεί και κατά το παρελθόν. Πολλοί άνθρωποι δεν κοιτάνε πια καθόλου τηλεόραση, ε, κοιτάνε μόνο βίντεο on demand, αυτά δηλαδή που δεν προβάλλονται από, μια, από ένα κλασικό ραδιοφωνικό τηλεοπτικό σταθμό. Ως εκ τούτου ε, στην ε, επανεξέταση αυτού του κανονισμού κάποια μεταγενέστερη στιγμή ε, θα πρέπει να σκεφτούμε το τι ισχύει με το video on demand σε αυτή την πλατφόρμα και να μην επεκταθεί και εκεί η αρχή της χώρας προέλευσης. Κυρία Λαγκρίπ, ε, γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχουμε την ακρόαση στις 5. Πρόεδρε, Ευχαριστώ στον εισηγητή που παρουσίασε. Δύο λόγια μόνο για τα δύο βασικά άρθρα που είναι στην κάρδια του κανονισμού. Στο άρθρο 2 προτείνεται η επέκταση της αρχής της χώρας προέλευσης στις επικουρικές υπηρεσίες των σταθμών εκπομπής μέσω διαδικτύου. Θα λέγει κανείς ότι η επέκταση αυτής της αρχής, η εφαρμογή της αρχής προελεύσης δηλαδή, θα μπορούσε να έχει το πλεονέκτημα της διευρυμένης πρόσβασης σε περιεχόμενο για τους Ευρωπαίους. Εγώ θεωρώ δυστυχώς ότι θα μπορούσε να έχει, θα έχει μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Περιχαρακώνουμε λοιπόν την πρόσβαση σε εθνικό επίπεδο. Έτσι θα αυξηθεί το κόστος των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Ανατρέπουμε λοιπόν μια κατάσταση, ένα σύστημα το οποίο εν γέννη βασίζεται σε κοινώς αποδεκτές αρχές. Την προβλέψιμη, σταθερή, χρέωση κλπ. Είναι η αρχή, οι αρχές αν θέλετε πάνω στους οποίους βασίζεται ένα ολόκληρο σύστημα και το οποίο ήδη λειτουργεί. Σήμερα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεργεί έρευνα όσον αφορά τις ρήτρε ορισμένων συμβάσεων που επιβάλλουν τα κανάλια. Το αποτέλεσμα φυσικά αυτής της έρευνας θα έχει επιπτώσεις στην οδό που θα ακολουθήσουμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε το πόρισμα αυτής της έρευνας. Θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παράλληλα επί του άρθρου 2 έτσι ώστε να μην αποσταθεροποιήσουμε ένα ήδη λειτουργούν σύστημα. Για το ΕΛΚ αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προτείνει μια αναδιατύπωση του άρθρου 2, αλλιώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεύτερο σημαντικό άρθρο είναι το άρθρο 3, το οποίο άπτεται περισσότερο των ε, τεχνικών μάλλον προσαρμογών που αφορούν ε, την οδηγία κάψα του 1993, όπου επεκτείνεται η υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στην περίπτωση ταυτόχρονης αναμετάδοσης μέσω κλειστών κυκλωμάτων μετάδοσης. Ενδιαφέρον διευκρινίζουμε λίγο την κατάσταση εδώ και κάποιες νομικές πτυχές όσον αφορά την πληρωμή, την αμοιβή μάλλον για δικαιώματα. Θα δούμε τώρα κάποιες συγκεκριμένες διατάσεις, αλλά για να μην μακρηγορώ, στο άρθρο 3 είμαστε και εδώ έχουμε μια πρόταση, η οποία νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα. Θα δούμε που θα πάει η συζήτηση από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χάνιμπολ, παρακαλώ, είστε σύντομοι. Πρόεδρε, για την επενεθνικοποίηση των αγορών, τη γεωγραφική περιχαράκωση, για όσους ε, γνωρίζουν τον τομέα, τον οπτικό, ακουστικό, για τους παραγωγούς προγραμμάτων, η δυνατότητα πώλησης υπάρχει, ε, έτσι μπορούν να επενδύσουν σε περιεχόμενο, Όμως, φοβούμαι ότι αν προχωρήσουμε έτσι, αν απαγορεύσουμε, αν δυσκολεύσουμε δηλαδή τις επενδύσεις, θα χάσουμε μερικά προγράμματα πολύ ψηλή ποιότητας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να επενδύσουν σε περιεχόμενο υψηλή ποιότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να προστατεύσουμε αυτό το περιεχόμενο υψηλή ποιότητα στην Ευρώπη. Προσωπικώ, ε, επειδή με ενδιαφέρουν και οι αγγλικέ παραγωγέ παραγωγές στην αγγλική γλώσσα εάν απελευθερώσουμε εντελώ την αγορά φοβούμε ότι θα χάσουμε το ευρωπαϊκό περιεχόμενο, οι Αμερικανοί θα εισβάλλουν, θα αγοράζουν άδειε, θα αγοράζουν τα πάντα και μακροπρόθεσμα θα είμαστε χαμένοι. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Έχει σημασία να μπορούμε να ακούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να ακούμε και να βλέπουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε και όχι να περιοριστούμε στην αγγλική γλώσσα. Και κάτι άλλο για το geo-blocking, την γεωγραφική περιχαράκωση, την απαγόρευση που επιβάλλουν ε, κάποιοι παραγωγοί. Ε, οι επιχειρήσεις αυτές χρηματοδοτούνται με παράξενο τρόπο. Έτσι εξασφαλίζουν τα έσοδά τους. Αυτό μπορεί να επηρεάζει και οι βρετανικές επιχειρήσεις, όχι το BBC. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε στο να καταργήσουμε το geo-blocking, αλλά σίγουρα υπάρχουν θέματα εδώ που μας ανησυχούν. Να το δούμε. Και υπάρχει και η περίπτωση CJU ε, Sky, τις επιπτώσει τι οποίε πρέπει να δούμε και εμεί εδώ. Κύριε Ροζιέρ, ξύδουμε παρακαλώ. Όσο πιο γρήγορα μπορώ, Πρόεδρε, είμαι υπέρ τη προλαλήσεω σα. Εδώ έχουμε μία σειρά υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου που βασίζεται σε μια μορφή αλληλεγγύης, αν θέλετε, μεταξύ παραγωγών, καναλιών, καλλιτεχνών κλπ. Εμείς τι θέλουμε. Για τους δορυφόρους υπάρχει η αρχή της χώρας ε, πρόλευσης, Όμως, οι επικουρικές υπηρεσίες γίνονται όλο και λιγότερο επικουρικές. Δεν πρόκειται για περιφερειακό πλέον φαινόμενο. Η κατάσταση αλλάζει. Η οικονομία αλλάζει. Η διαπραγμάτευση περί δικαιωμάτων, όπως είπε και η Μαρή, αλλάζει και αυτή. Πρέπει να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης ενός έργου. Τα προγράμματα δεν δημιουργούνται εκ του μηδενός. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους δημιουργούς. Και σχετικοί μηχανισμοί ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει να σταθούμε στο πλάι των δημιουργών. Η δημιουργία σημαίνει μία φορά προφανώς σε μια συγκεκριμένη χώρα και από εκεί πέρα θέλουμε να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό. Εν δεν κατάλαβα την πρόταση της Κομισιόν. Έχουμε βεβαίως τις κρατικές τηλεοράσεις που παρέχουν περιεχόμενο ενημέρωση κλπ. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των καναλιών, παραγωγών κλπ. είναι ικανοποιημένοι από την παρούσα κατάσταση και δεν θέλουν να αλλάξουν με τίποτα. Γιατί λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα, αν το σύστημα λειτουργεί. Και όπως είπε η κυρία Λαγκρίπ, όσον αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα στις ενσύρματες αναμεταδόσεις. Γιατί υποχρεωτική λοιπόν συλλογική διαχείριση στον τομέα αυτών. Δεν ξέρω. Ίσως γιατί όχι. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα τα οποία διευκολύνουν την διασυνοριακή αναμετάδοση με την προϋπόθεση βεβαίω ότι όλοι αμείβονται δίκαια. Πάντως η αρχή της χώρας προέλευσης δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται πλέον σε κάποια πραγματικότητα. Δεν λειτουργεί πλέον έτσι ο οπτικο-ακουστικός τομέας. Ευχαριστώ. Μήπως η Κομισιόν έχει σύντομο μήνυμα για μας. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Γιώτα να από την Γενική Διεύθυνση Connect. Να σας πω δύο λόγια. Μιας δεν έχουμε χρόνο, θα τα πω γρήγορα. συνολική πρόσβαση σε προγράμματα. Για τους στόχους της Κομισιόν να μιλήσω και αποφορούν διάφορες ερωτήσεις. Η συγγήτρια τα, προ... τα παρουσίασε σωστά. Να προσθέσω μόνο το εξή. Πριν χρόνια είχαμε στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση για διασυνορικές υπηρεσίες και πρόσβαση. Πανευρωπαϊκά, όχι μόνο από κάποιες μειονότητες γλωσσικές ή εθνοτικές. Και αυτό έως αφορά τους Ευρωπαίους φορείς τηλεπικοινωνιών. Σήμερα θα ήταν καλό λοιπόν να υπάρχει ευρεία πρόσβαση για τους Ευρωπαίους πολίτες και για να πετύχουμε αυτό το στόχο στην πρόταση έχουμε ένα μηχανισμό διευκόλυνσης όχι υποχρεωτικό διευκόλυνσης που θα διευκολύνει δηλαδή τους μεταδότες να φτιάξουν προγράμματα κάθε φύσης Όταν κάνουμε αξιολόγηση αντικτύπου, βλέπουμε ότι αυτό το περιεχόμενο γεμπλοκάρεται. Αλλά για το περιεχόμενο, νομίζω υπάρχει ελευθερία. Δηλαδή, δεν επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες από οργανισμού που παράγουν προγράμματα. Και πρέπει να δούμε ακριβώ και το πώ ε, γίνεται η παραγωγή και χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων στην Ευρώπη. Επειδή λοιπόν αυτά είναι μέτρα διευκόλυνση και αφήνουν δεκατική ευχαίρεια και ελευθερία, δεν ε, ασχολούμαστε, δεν καλύπτουμε τι μαυροπαϊκέ άδειε γιατί οι επιχειρήσει είναι ελεύθερε να λάβουν αποφάσεις σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών τους. κάποιοι μέλη τη Επιτροπή σα αναφέρθηκαν σε κάποιες υποθέσεις ανταγωνισμού. Να κάνω κάποια σχόλια. Να τονίσουμε ότι εξετάσουμε συγκεκριμένα δεδομένα και μέτρα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην τα ανακατέψουμε περιτά. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα δεδομένα και που αφορούν συγκεκριμένους στόχους, ώστε ακριβώς να μην διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά έχουμε λοιπόν ρυθμιστικές διατάξεις όπως τώρα προτείνεται, εμείς δεν αφισβητούμε την πρακτική του αποκλειστικού παρόχου ή της περιφερειακής άδεια. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε το ότι ο, η νομοθεσία ανταγωνιστικότητας ανταγωνισμού συγγνώμη λαμβάνει υπόψη σε συγκεκριμένε συνθήκε που επικρατούν στην κάθε αγορά όταν ξεκινούν νέες μορφές υπηρεσιών. Δηλαδή, υπάρχει ελευθερία να αποτιμήσουμε το πώς ακριβώς με μονομένα τηλεοπτικά προϊόντα χρηματοδοτούνται. Και αυτό το το κάνουμε ελέγχοντας συγκεκριμένα στοιχεία που τα συνοδεύουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση θα έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και τους καταναλωτές, χωρίς βεβαίως να θίξει κάποιες φανατικότητες που ισχύουν στην αγορά και τους κανόνες της αγοράς. Και προσβλέπουμε σε περισσότερες συζητήσεις η συνεργασία με το Κοινοβούλιο σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο. Σημείο 20. Κοινή ακρόαση. Επιτροπών απασχόλησης και τζούρι. Η κυρία Μαρίτα Ούσκο και αντιπρόεδρος θα μιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά να σας πω ότι η εκρόαση θα αφορά το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων. Και μιας και έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά, και να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη της Apple θα ζητήσω από τον άλφα να μας πει αν θέλει να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Ναι, να πω και εγώ δύο λόγια λέει η Αντιπρόεδρος. Καταρχάς ευχαριστώ που μας καλέσατε σημαντικό να συνεργαζόμαστε ως επιτροπές συνδυάζουμε για ώρες συνδυάσαμε για ώρες και συζητήσαμε τα θέματα απασχόλησης προσωρινής και ανασφαλούς απασχόλησης και το πώς θα αλλάξουμε την αγορά εργασίας ώστε ο κόσμος να βρει δουλειά, να έχει εισόδημα και να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του. Αυτό κάνουμε και θέλουμε συμμάχους αυτό. Και χαιρόμαστε που η Επιτροπή Γιούρι θέλει να συμμαχίσει με μας. και να συζητεί το θέμα κοινωνικό και ελόγιων επιχειρήσεων. Γιατί πολλοί βουλευτέ εδώ έχουν εμπειρία για το πόσο καρποφόρα είναι αυτή η προσπάθεια στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε και χαιρόμαστε ξεκινάμε τώρα, ακούγοντας τις δικές σας θέσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Έχουμε και μία intergroup, ομάδα στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί εταίροι που μπορούν να βοηθήσουν. Και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, ξαναλέω. και λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ώστε να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Ε, ε, μου ζήτησαν να κάνουμε διάλειμμα ενό λεπτού λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων στις καμπίνες διερμηνίας. Να σου δώσουμε λοιπόν κάποια δευτερόλεπτα για να το λύσουμε.